Συνάδελφοι, νομίζω θα ξεκινήσω αμέσως. Σε όλες τις επιτροπές προσφάτως έχουμε προβλήματα με την προσέλευση των συναδέλφων και από ό,τι μαθαίνω λόγω των εκλογών θα χειροτερέψουν και τα πράγματα. Ε, να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Όπως ξέρετε θα μεταδοθεί και στο διαδίκτυο. Να ξεκινήσω με το σημείο 1 της ημερήσιας διάταξης που είναι η έγκριση αυτής έχει διανεμηθεί από τις 15 Νοεμβρίου. Και να σας ενημερώσω ότι πριν τις ψηφοφορίες θα αποφασίσουμε αν θα γίνουν αλλαγές στην ημερήσια διάταξη ή όχι. Ε, για την ώρα δεν έχω άλλες, άλλα αιτήματα για αλλαγές, οπότε γκρίνεται η ημερήσια διάταξη και θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι θα ψηφίσουμε για τις εκθέσεις Λάινεν και Τόμ βάσει του, του άρθρου 55 και για τη διαφάνεια των κοινωνικών συζητήσεων στα προπαρασκευαστικά σώματα του Συμβουλίου. Αυτό θα γίνει αύριο 9 με 9.30. Την χρονοθερίδα της κοινή συνεδριασής μας με την ΠΕΤΗ. Παρακαλώ όσοι βρίσκεστε στο Κοινοβούλιο ή στις Βρυξέλλες, ελάτε αύριο σε αυτή τη συνεδρίαση για να ψηφίσουμε. Δεύτερη ανακοίνωση. Πρωτοβουλίε των πολιτών. Είχαμε δύο πολύ καλούς γύρους τριμερούς διαλόγου. Εξαιρετική τεχνική δουλειά. Προχωρήσαμε σημαντικά με αρκετές πιθανότητες να βελτιώσουμε και να οδηγηθούμε σε αίσιο πέρας επί Αυστριακής Προεδρίας. Υπάρχει βέβαια και υπάρχουν και οι πικάντικες λεπτομέρειες. Το Συμβούλιο στο Στρασβούργο ε, μας ανακοίνωσε ότι θα πρέπει να ξαναπάει στα κράτη-μέλη και να ζητήσει να κοιτάξουν κάποιες τροπολογίες για κάποιους προβληματικούς τομείς κυρίως για το όριο ηλικία, αυτών που είναι επιλέξιμοι να συμμετέχουν σε πρωτοβουλία πολιτών. Όπως ξέρετε, το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή θέλαμε να πάμε στα 16 έτη ηλικία. Και κάτι άλλο που συζητιέται στο Συμβούλιο είναι η ατομική συλλογή δεδομένων ε, στο διαδίκτυο. Και μετά και ο νέος κύκλος ζωής των πρωτοβουλίων των πολιτών αλλά με τη συζήτηση που θα έχουμε με τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα θα μπορέσουμε να το ολοκληρώσουμε αυτό. Πολύ σύντομα θα κοιτάξω να σας ενημερώσω καλύτερα την επόμενη φορά στην Κόζακ. Σάββατο, Κυριακή, μάλλον Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη στη Βιέννη συμμετείχαμε και εμείς με πολλά σημαντικά ζητήματα προς συζήτηση. Το Brexit προφανώς, θέματα της Αυστριακής Προεδρίας, την ενέργεια και το κλίμα, το ρόλο των πολιτών στην ευρωπαϊκή πορεία ολοκλήρωσης και την ανάγκη να έρθουμε πιο κοντά στους πολίτες. Πολύ καλές συζητήσεις με τα Εθνικά Κοινοβούλια και την ε, συμμετοχή των Εθνικών Βουλευτών. Αυτά από δική μου πλευράς ως προς τις ανακοινώσεις. Τζόρτζ. Ευχαριστώ. Ναι, απλώ μια επιπλέον παρατήρηση για, την πρωτοβουλία, για τι πρωτοβουλίε των πολιτών. Νομίζω ότι την επόμενη εβδομάδα έχουμε τρίτο γύρο τριμερού διαλόγου, έτσι. Εκεί θα ενημερώσουμε για τα εκκρεμή ζητήματα, θα κοιτάξουμε τα εκκρεμή ζητήματα. Εάν καλά κατάλαβα και αν όλα πάνε καλά, η Αυστριακή Προεδρία θα έχει νέα εντολή για να δούμε τα εναπομείνοντα ζητήματα. Θα θέλαμε να έχουμε ολοκληρώσει, αν γίνεται, μέχρι τα Χριστούγεννα. Φαντάζομαι ότι και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπάρχει αυτή η διάθεση να ολοκληρωθεί εγκαίρω το θέμα. Ο νέο κανονισμό, το νέο σύστημα να λειτουργήσει από την 1η Ιανουαρίου του 2020. Ευχαριστώ πολύ για αυτά τα σχόλια. Πάμε στο σημείο 3 τώρα, έγκριση των πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων, 25 Απριλίου, τα πρακτικά είναι διαθέσιμα και ως ήθιστε, εάν δεν υπάρξουν αντιρρήσεις μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, θα θεωρηθούν εγκεκριμένα. Επίσης, ενημερώνομαι ότι αλλάζουμε τη σειρά. Ο κύριος Μέσερ Σμιτ, που θα παρουσίαζε πρώτος τις τροπολογίες στην έκθεσή του, για το εσωτερικό καταστατικό του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι ακόμη εδώ, οπότε θα συζητήσουμε με την κυρία Μπρέσο για την πολύ ουσιαστική έκθεσή της, για τον ε, δημοκρατικό έλεγχο του Κοινοβουλίου στο έργο της Επιτροπής. Μπρέσο, ευχαριστώ Πρόεδρο. Πρόεδρε, θα μιλήσω γαλλικά. Ε, όπως γνωρίζετε, έχουμε μία έκθεση για τον πολιτικό έλεγχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θεωρώ ότι πρόκειται για κεντρικό σημασία ε, θέμα σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία πολύ έχει εξελιχθεί τα δέκα τελευταία χρόνια. Η θεσμική δομή επίσης ε, έχει τροποποιηθεί και εξελιχθεί ε, λόγω και εξαιτία των πολλών κρίσεων, εξελίξεων, στοιχείων κλπ. Τα τελευταία χρόνια είχαμε πολλά νέα στοιχεία. Πρώτον, συνθήκη Λισαβόνας, νέα θεσμική δομή. Ε, δεύτερον, η ιδέα του Spitzenkandidat, δηλαδή η άμεση εκλογή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βάσει των αποτελεσμάτων των ευρωπαϊκών εκλογών, πράγμα που σημαίνει ή θα έπρεπε να σημαίνει ε, πολιτικό έλεγχο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τρίτο, η ε, ε, ε, πρόσφατη μη κωδικοποιημένη τροποποίηση των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου που έγινε κατά κάποιο τρόπο συν νομοθέτης και συν εκτελεστική εξουσία. Εμείς ε, θα πρέπει οπωσδήποτε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, να θεσμοθετήσουμε τις ε, σχέσεις μας με τον, τον νομοθετικό και εκτελεστικό σκέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να διατηρήσουμε την παραδοσιακή μορφή των κοινοβουλίων αλλά και να προωθήσουμε τη θέση μας ως συνομοθέτη. Οι στόχοι της εκθέσεώς μου είναι οι εξής. Πρώτον, να κάνω έναν ε, απολογισμό του συνόλου των στοιχείων και αφετέρου ε, να κάνουν συστάσεις ε, ή ε, οποιασδήποτε τροποποιήσεις έτσι ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση. Έχουν γίνει, έχει γίνει εργασία πολλών μηνών. Είχαμε και στις 10 Οκτωβρίου τον κύριο Ολιβιέ Κωστά και την κυρία Πουλτσέβα που μας, με τις οποίους συζητήσαμε το θέμα αυτό. Η γραμματεία έχει βοηθήσει ιδιαίτερα Κυρίω κυρίως η κυρία Τομπαλόβα, την οποία θα ήθελα να ευχαριστήσω και θα ήθελα βεβαίως να ευχαριστήσω και τις υπηρεσίες έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ε, εξαντλητική και ε, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εργασία τους. Δεν ξέρω αν την έχετε δει ήδη, να τη δείτε γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Τρεις είναι οι άξονες προβληματισμούς αυτήν την ε, έκθεση η οποία όπως βλέπετε είναι αρκετά πλούσια. Άρα θα πρέπει οπωσδήποτε ε, να συμπτύξω κάπως ε, τις ιδέες. Τρεις άξονες έλεγα. Ε, πρώτον, να εκμεταλλευτούμε όσο γίνεται περισσότερο τις δυνατότητες που δίνονται από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Το πρώτο πρόβλημα όμως που προκύπτει είναι ότι η συνθήκη δεν δίνει σαφή ορισμό ε, για τον τρόπο με τον οποίο ε, και ποιος μάλλον εκτελεί ε, τις εκτελεστικές εξουσίες και τις νομοθετικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δίνονται και περιθώρια ε, σχέσεις και με τις περιφέρειες, κυρίως αυτές που έχουν και νομοθετικές εξουσίες. Επίσης έχουμε την multi-level governance που καθιστά δύσκολο τον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επίσης σε εθνικό επίπεδο ή περιφερειακό μερικές φορές επίπεδο ή ε, αρμόδιοι για τον έλεγχο δεν έχουν ε, τις απαραίτητες ικανότητες γνώσης για αυτόν τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, πράγμα που καθιστά την όλη ε, κατάσταση πολύ πιο περίπλοκη. Δεν ξέρουμε δηλαδή πώς γίνεται η εκτέλεση στο τέλος. Ο έλεγχος του Κοινοβουλίου, έτσι όπως αναφέρεται στο άρθρο 14 της Συνθήκης Λειτουργίας, ε, μπορεί να ασκηθεί ε, μόνο εάν ξέρουμε ποιος ακριβώς ασκεί τις εκτελεστικές εξουσίες. Ένα άλλο σημείο είναι το εξής. Στα πλαίσια της συνθήκης του Λισα, της ε, υπάρχουν, πρέπει να εισαχθούν στοιχεία τα οποία δεν μπορούν να ελέγχονται από το Κοινοβούλιο, μάλλον έχουν εισαχθεί το Fiscal Compact ας πούμε. Ε, εδώ γίνεται μια ολόκληρη συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να ενταχθούν στη συνθήκη της ε, Λισαβόνας αυτά τα στοιχεία. Άρα μέχρι να ενταχθούν δεν μπορούν να ελεγχθούν. Επίσης, το άρθρο 225 ε, μας δίνει τη δυνατότητα να ε, υποβάλουμε αιτήματα στην Κομισιόν. Μονάχα μία όμως από τις 7 προτάσεις ε, πήρε πράσινο φως από την Κομισιόν. Αυτή η κατάσταση θα πρέπει να εξελιχθεί. Θα πρέπει η Κομισιόν να βλέπει με θετικό μάτι τις προτάσεις αυτές, τις οποίες δίνει στο Κοινοβούλιο η συνθήκη άλλος άξονας, ο έλεγχος που δεν είναι ικανοποιητικό για το Κοινοβούλιο. Όπως ξέρετε, η διαδικασία του Spitzenkandidaten έχει προκαλέσει πολιτικοποίηση της Κομισιόν, αλλά δεν έχει ε, προκαλέσει και αλλαγή ε, των συνθήκων, γιατί δεν προβλέπεται από τις συνθήκες. Θα ήταν ε, πολύ καλύτερο να ανοίξουμε τον δρόμο προς ε, μεμονωμένο έλεγχο των, ε, του Κοινοβουλίου ε, για τους μεμονωμένους επιτρόπους. Αυτή τη στιγμή οι απαραίτητες προ... πλειοψηφίες, ας πούμε δύο τρίτα για πρόταση μομφής, επειδή δεν μπορούν να επιτευχθούν, καθιστούν την όλη διαδικασία μη πραγματοποιήσιμη. Ε, δεύτερον, ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να ξεκαθαριστούν οι, ε, λειτουργίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξουν και οι πρακτικές ακόμα και αυτές του Κοινοβουλίου. Δηλαδή, οι τα ε, θέματα τα οποία μπορεί να ε, γίνονται δεκτά βάσει του άρθρου 129 η ενίσχυση των ισχνών ικανοτήτων του Κοινοβουλίου για ε, έλεγχο των κατεξουσιοδότηση πράξεων. οπωσδήποτε θα πρέπει να γίνει πιο κοινοβουλευτική η Ευρώπη έτσι ώστε να καλυφθεί και το δημοκρατικό κενό και έλλειμμα και έτσι ώστε να ασκηθεί ε, η ε, νομοθετική εξουσία και οι δημοκρατικές διαδικασίες με έναν ε, καλύτερο και πιο αποτελεσματικό τρόπο Βεβαίω Βεβαίως εδώ χρειάζεται και αλλαγή των συνθήκων, αναθεώρηση των συνθήκων, αλλά θα μπορούσε να γίνουν και κάποιες συμφωνίες όπου θα προβλέπονται κάποια στοιχεία μέτρα ελέγχου. Επίσης, θα πρέπει να αναγνωριστεί η ε, η δυνατότητα του Κοινοβουλίου να ελέγχει το εκτελεστικό τμήμα μέσω ας πούμε ε, των ε, ακροάσεων των ε, επιτρόπων ή ακόμα και μέσω ακροάσεων των υψηλών αξιωματούχων υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που οπωσδήποτε έχουν αρμοδιότητες περίπου αντίστοιχες με τους υφυπουργούς των κυβερνήσεων. Επίσης, Έχουμε μεγάλο πρόβλημα εμείς πάντα να ε, νομοθετήσουμε τις επιτροπές ε, έρευνας, έστω και αν ε, θα έπρεπε να είναι διαφορετική η κατάσταση. Επίσης, γίνονται διάφορες συστάσεις, γίνονται πολλές προτάσεις, οι οποίες ε, δίνουν κάποια ε, νέα στοιχεία. Κυρίως ε, λέμε ότι θα πρέπει οπωσδήποτε ο επιμερισμός των ευθυνών για, την, για τον έλεγχο θα πρέπει να είναι σαφέστερος. Επίσης αυτά τα νέα στοιχεία της πολιτικοποίησης της Κομισιόν από την Λισαβόνα και μετά θα πρέπει να μας δώσει κάποια, κάποιες επιπλέον δυνατότητες. Όσοι διαβάσατε ε, την έκθεση θα έχετε καταλάβει ότι είναι πάρα πολύ σημαντική έκθεση γιατί θα δηλώσει και την ε, θέση μας ε, σαν Κοινοβουλίου και θα ολοκληρωθεί και η θητεία με ικανοποιητικό τρόπο αλλά ταυτόχρονα θα δώσουμε και κάποιες ε, κάποια θετικά στοιχεία και στους ε, διαδόχους μας μετά από τις εκλογές του 2019. Ελπίζω ότι θα έχετε το χρόνο να το διαβάσετε. Σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας και για τις παρατηρήσεις σας. Η ημερομηνία κατάθεση των τροπολογιών θα οριστεί, αλλά μέχρι τότε εκ των προτέρων σας ευχαριστώ για τις συμβολές που θα στείλετε. Πρόεδρος, ευχαριστώ Μερσέντες. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος από τους κοιόδης να μιλήσει. Ο Έλμαρ δεν είναι εδώ. Ο κύριος Μέσο Σμιτ δεν είναι εδώ. Would Πασκάλ, που είσαι εδώ, θες να πεις κάτι. Ναι. Ε, να απαντήσω κι εγώ γαλλικά, μια και η Mercedes ε, μίλησε στα γαλλικά, να πω ότι την υποστηρίζω ε, ολόθερμα και της έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Και εγώ να μιλήσω στα γαλλικά, λέει ο κύριο Κόρμπιν. Είναι εξαιρετική η έκθεση, πάρα πολύ ωραία, μπράβο σας και έβγε σα. Αλλά τώρα θα τα πω γαλλικά, λέει ο κύριο Γιολάιν. <clears throat> Ja, der Bericht äh, äh, äh, zeigt sehr schön. Βλέπουμε λοιπόν ε, με απόλυτη σαφήνεια πως το Κοινοβούλιο με πολύ μεγάλο κόπο απέκτησε τις αρμοδιότητές του. Πάρα πολλά από αυτά που έχουμε σήμερα ως αρμοδιότητες ελέγχου δεν υπάρχουν στις συνθήκες και νομίζω ότι ε, πολλές φορές μπορέσαμε να διεκδικήσουμε δικαιώματα για τις πολίτες ε, παρά τις αντιστάσεις και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τις εθνικές κυβερνήσεις. Νομίζω λοιπόν ότι ανεξάρτητα από την νομική βάση ε, έχουμε περισσότερες αρμοδιότητες ελέγχου από πολλά εθνικά κοινοβούλια στα κράτη-μέλη. Ε, αυτό είναι τελείως διαφορετικό. Η Mercedes έθεσε τον δάκτυλο σε έναν ήλο που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ήλος αυτός είναι ότι ε, δεν έχει οριστεί ακριβώς σε ποια είναι η εκτελεστική εξουσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε πολλές εκτελεστικές εξουσίες. Το καλύτερο είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει εκτελεστική εξουσία το καλύτερο λοιπόν από όλα ε, θα είναι το ε, Συμβούλιο να αναλαμβάνει νομοθετικές πρωτοβουλίες. Πιστεύω λοιπόν ότι η προσπάθειά μας προς το θέμα είναι ότι θα πρέπει να προβάλλουμε τις ε, εκτελεστικές αρμοδιότητες με την έννοια ότι η Επιτροπή οφείλει στον τομέα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης να έχει περισσότερες αρμοδιότητες και να ελέγχεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όσον αφορά τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παραδοσιακά έχουμε το, την ψήφο δυσπιστίας ε, και αυτό έχει απομείνει από το παρελθόν. Βέβαια, μόνο συλλογικά μπορούμε να εκφράσουμε τη δυσπιστία μας έναντι της Κομισιόν, αλλά όχι έναντι ενός και μόνο επιτρόπου. Και αυτό είναι πλέον απαρχαιωμένο. Έχει έρθει η στιγμή έτσι ώστε να μπορούμε να αναζητάμε ευθύνες, ε, από ένα και μόνο άτομο ε, και έναν και μόνο επίτροπο και να μην χρειαστεί να χρησιμοποιούμε πυρηνικά όπλα κατά της Κομισιόν, δηλαδή να είμαστε αναγκασμένοι να την αποπέμψουμε στο σύνολό της. Ε, θέλω να σας πω ότι ε, μην δεν είμαστε ευχαριστημένοι με το ότι δεν έχουμε το δικαίωμα της διεξαγωγής ερευνών. Και αυτό είναι σκάνδαλο το ότι το Συμβούλιο δεν μας δίνει αυτή την αρμοδιότητα στα, ε, στις διάφορες διαρροές, ε, Panama Papers, Lux Papers. Είδαμε πόσο χρήσιμο θα ήταν οι πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορούν να προσκαλούν μάρτυρες για να καταθέσουν ε, που πολλές φορές δεν το κάνουν ε, εθελοντικά γιατί δεν θέλουν να εκτεθούν σε ερωτήσεις. Ε, θα ήθελα να αφαιρθώ και στο νομοθετικό δικαίωμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το μονοπόλιο για την ανάληψη πρωτοβουλειών. Μετά από πολλές δεκαετίες αυτό είναι απαρχαιωμένο. Το Κοινοβούλιο πρέπει να έχει το δικαίωμα της ανάληψης πρωτοβουλειών. Και εμείς απλά χρησιμοποιούμε ένα δεκανίκι ε, δηλαδή ε, παρακαλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εφαρμόζει τις ε, νομοθετικές μας ιδέες. Βεβαίως, τι να κάνουμε, θα βολευτούμε με αυτό το δεκανίκι μέχρι να υπάρξει μια νέα συνθήκη, αλλά το δικαίωμα διεξαγωγής ερευνών και το νομοθετικό δικαίωμα είναι, αναφέρεται δικαιώματα πρωτοβουλίου και αυτά είναι τα επόμενα που πρέπει να διεκδικήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Ο Γιολάινερ μόλις τώρα ανέφερε πως ε, πολλές από τις αρμοδιότητες που έχουμε ε, απλά ήταν το αποτέλεσμα διεκδικήσεών μας ε, στη διάρκεια των ετών. Και ας πούμε, δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη στη συνθήκη για το ότι θα πρέπει να προηγούνται ακροάσει πριν διοριστούν οι επιτροποί. Αυτό όμω το πετύχαμε και τώρα είναι ένα σύστημα που λειτουργεί αρκετά καλά στο κείμενο της αιτιολόγησης ε, βλέπω εκεί αναφέρονται τρία παραδείγματα ε, επιτρόπων που μετά από αρνητική ακρόση αναγκάστηκαν να αποσύρουν την υποψήφιά τους. Υπάρχει και μία ε, τέταρτη περίπτωση, αλλά εν πάση περιπτώσει, εκτός από το ότι αναγκάστηκαν να αποσύρουν την υποψηφιότητά τους, υπήρξαν και περιπτώσεις όπου μερικοί αναγκάστηκαν να αλλάξουν χαρτοφυλάκιο. Και αυτό ως αποτέλεσμα της ακρόασης. Όσον αφορά τώρα το θέμα της εκτελεστικής εξουσίας ή των εκτελεστικών εξουσιών, νομίζω ότι ε, όλοι γνωρίζουμε ότι η εκτελεστική εξουσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι αλήθεια ότι το Συμβούλιο μερικές φορές μπορεί να επιφυλάξει κάποια δικαιώματα στον εαυτό του, αλλά αυτό είναι μία εξαίρεση στον κανόνα. Και κατά κανόνα εμείς δεν δίνουμε εκτελεστικές εξουσίες στο Συμβούλιο. Το Συμβούλιο πολύ συχνά αντιμετωπίζεται ως εκτελεστική εξουσία, κυρίως σε, σε γαλλόφωνες χώρες, λόγω του Conseil de Ministres. Είναι ε, σαν ε, να είναι το, ε, ο εκτελεστικός βραχίωνας. Βλέπετε λοιπόν ότι και τα δικά μου τα γαλλικά μια χαρά είναι. Mm. Και στην Ιταλία ισχύει αυτό, ε, όπου υπάρχει το Conseil de Ministres, ε, δηλαδή αυτό ηχεί ως εκτελεστική εξουσία. Ενώ στα γερμανικά ε, η λέξη Rat υπενθυμίζει στους πολίτες ε, την κάτω βουλή, το Bundesrat, η βουλή που εκπροσωπεί τα κρατήδια. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχουν διαφορετικέ ερμηνείε και νομίζω ότι συμφέρει το Κοινοβούλιο να περιορίσει την άποψη ότι το Συμβούλιο είναι η εκτελεστική εξουσία. Το ίδιο ισχύει και για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Είναι ο φορέας εκείνος ε, που υποτίθεται ότι καθορίζει τις προτεραιότητες ε, και την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν βέβαια επικρατεί συνένεση. Όμως ε, δεν λαμβάνει αποφάσεις άμεσα σε αντίθεση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει το δικαίωμα να προτείνει νομοθετικό έργο ούτε να εφαρμόζει, να εκτελεί τον προϋπολογισμό. Πρώτα ο πρόεδρος Βαν ε, Ρομπό ήταν ο πρώτος ε, που είπε ότι είναι ένας ε, σταθμός παραγωγής ρεύματος που όμως δεν συνδέεται με το ηλεκτρικό δίκτυο και πρέπει να ακολουθήσουν πάντα και άλλοι θεσμοί στο πλαίσιο της κοινοτικής μεθόδου. Ως εκ τούτου μερικοί άνθρωποι λένε ότι είναι σαν να έχουμε έναν συλλογικό πρόεδρο της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το γαλλικό σύστημα, όπου έχουμε τον Πρωθυπουργό, αλλά έχουμε τον Πρόεδρο, έχουμε τον Πρωθυπουργό, την Κυβέρνηση και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι ένα ίδιος σε ένα ημιπροεδρικό σύστημα. Αυτά, αυτές οι συγκρίσεις δεν λειτουργούν βέβαια απόλυτα, αλλά νομίζω ότι έτσι αποκτά κανείς μια ιδέα ότι η πραγματική εκτελεστική εξουσία είναι η Επιτροπή. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει κάποιο ρόλο, αλλά ε, δεν είναι ότι έχει τη δυνατότητα να εφαρμόζει ε, προγράμματα. Ο κύριο Σέπλιν, ε, δεν θα σας βασανίσω με τα γαλλικά μου, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά για την έκθεση της Mercedes πρέπει να πω ότι πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Και στη δική μου την έκθεση ασχολήθηκα και εγώ με κάποιους από τους οργανισμούς που σύντομα θα συζητήσουμε. Σε σχέση με όσα υπογειώ υπάρχουν πολλές αρμοδιότητες ελέγχου. Απλώς δεν τις ασκούμε, διότι δεν έχουμε το δικαίωμα πρωτοβουλίας, οπότε δεν ενεργοποιούνται ποτέ. Και από τη δουλειά μας με τις πρωτοβουλίες των πολιτών καταλήγω στο συμπέρασμα ότι δεν θα αφήσει ποτέ το δικαίωμα πρωτοβουλίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα το Κοινοβούλιο. Μπορεί να συζητά, έχει τη δυνατότητα να ασκεί δημοκρατικό έλεγχο και να δυσκολεύει τη ζωή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως έχουμε κάνει στο παρελθόν με πολλά θέματα συγκεκριμένα αναλόγως με το χαρτοφυλάκιο κάθε φορά ε, το θέμα είναι η πρώτη μου φορά στα 15 χρόνια που βλέπουμε Κάπω να αυξάνεται η δυνατότητα δημοκρατικού ελέγχου του Κοινοβουλίου, επειδή έχουμε λάβει και τη σχετική προβολή κτλ. Αλλά νομίζω εν τέλει η όλη διαχείριση του συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ξανασχεδιαστεί. Πρέπει να φτάσουμε στο ύψος των απαιτήσεων του 21ου αιώνα. και να υπάρχει η κατάλληλη προβολή για την κοινή γνώμη και βεβαίως να υπάρχει και το σύστημα που λειτουργεί όχι μόνο για λόγους διαφήμισης. Αλλά πραγματικά το πρόβλημα είναι ότι η συνθήκη που έχουμε στα χέρια μας ήδη αρχίζει να κλειδονίζεται. Ε, υπάρχουν τριγμοί δεν είναι κακή, αλλά πρέπει να έχουμε με πιο επιτυχημένη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και οι κυβερνήσεις νομίζω θέλουν, ε, από ό,τι τώρα συμβαίνει. Ευχαριστούμε ο κύριος Βίλαντ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για, αυτή, αυτό το πολύ ενδιαφέρον σχέδιο της έκθεσης ε, και θέλω μόνο να κάνω δύο προτάσεις. Νομίζω πρώτον ότι στην έκθεση αυτή ως ε, κοινοβούλιο μπορούμε να περιγράψουμε περισσότερα πράγματα. Μπορούμε, παραδείγματο χάρη, να περιγράψουμε πόσο επιτυχημένη ήταν η όλη διαδρομή μέχρι σήμερα. Η τη τελική ανάλυση, η έκθεση θα ψηφιστεί λίγο πριν από τις ευρωεκλογέ. Και εφόσον υπάρχει κάποια κοινή γνώμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να τι εξηγήσουμε από πού προερχόμεθα. Και θα σας αναφέρω δύο πράγματα. Για πρώτη φορά θα έχουμε τη δυνατότητα να ε, υποβάλει υποψηφιότητα ένας επίτροπος ε, και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό είναι κάτι ε, που δεν είναι αυτονόητο. Ε, μέχρι τώρα οι επίτροποι που φοβόντουσαν ότι θα επανεκλογούν, τι έκαναν. Κατέθεσαν παρέτηση λίγο πριν τις εκλογές και μετά εμφανίζονταν εκ νέου Ω υποψήφοι. Τώρα για πρώτη φορά ένας επίτροπος μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Από την εποχή του Μπαρόζο για πρώτη φορά ο πρόεδρος της Επιτροπής ε, για την κατάσταση της ε, Ένωσης όχι μόνο δεν έκατσε τη θέση του και δεν σηκώθηκε, αλλά μπήκε και στο κέντρο του Κοινοβουλίου, στην αίθουσα δηλαδή. Και αυτό είναι κάτι το απόλυτα καινούριο. Δηλαδή μετατίθεται και καθαρά σωματικά και φυσικά η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Νομίζω λοιπόν ότι στην έκθεση αυτή υπάρχουν θέματα που μας αφορούν, που μπορούμε να βελτιωθούμε, πρέπει να τα περιγράψουμε καλύτερα. Εγώ δεν νομίζω ότι μέχρι τώρα τις ακροάσεις τις οργανώνουμε σωστά ε, υπάρχει ένα, μια πολυμορφία, υπάρχουν πάρα πολλά. Έχουμε πρόεδρους των επιτροπών οι οποίοι ε, έγραψαν μια επιστολή, οι οποίοι ε, άκουσαν ορισμένα πράγματα και έστειλαν την επιστολή, επιστολή, άλλοι πάλι ψήφισαν. Εγώ θεωρώ ότι η έκθεση θα πρέπει να εξυπηρετήσει εμά, Μόνοι μας δηλαδή να γράψουμε ορισμένα πράγματα για το πού μπορούμε να βελτιωθούμε. Κατά τα άλλα, δυστυχώς ε, μια παρατήρηση εκτός μικροφώνου. Ο κύριος Βίλαντ λέει, θέλω να πω με απόλυτη σαφήνεια ότι αυτή η έκθεση θα ψηφιστεί λίγο πριν από τις ευρωεκλογέ. και γι' αυτό θα έχουμε την ευκαιρία να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Και θέλω να πω ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τη δήλωση του κυρίου Βίμπερ ότι επιθυμεί να γίνει πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ως εκ τούτου κατά κάποιον τρόπο βοηθάει το Κοινοβούλιο και επικρατεί άποψη ότι όπου το θέλει το Κοινοβούλιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναλαμβάνει πρωτοβουλία. Επιμπαρόζω αυτό ε, το είχε απορρίψει ο κύριος Μπαρόζο. Είχε πει εμείς ε, θα εξετάζουμε τις ε, προτάσεις του Κοινοβουλίου. Ο κύριος Γιούνκερ είχε πει και εμείς θα τις εξετάζουμε. Και μετά από έξι μήνες είτε θα αναλάβουμε πρωτοβουλία είτε θα πρέπει να αιτιολογήσουμε γιατί δεν αναλαμβάνουμε πρωτοβουλία. Αλλά ο κύριος Βέιμπερ ως σπίτσαν καντιντάτ δήλωσε ήδη ότι θέλει να κάνει ένα βήμα πιο πέρα. Είναι λοιπόν μικρά τα βήματάκια που γίνονται αλλά θεωρώ ότι τα βήματάκια αυτά θα πρέπει να εμφανίζονται στην έκθεση ως ένα φύγημα Πώ Πώς δηλαδή έχει αλλάξει η κατάσταση. Και τέλος πιστεύω ότι η έκθεση ναι μεν αναφέρεται στην ε, Κομισιόν αλλά και στο Συμβούλιο και αυτά τα είπαν ήδη οι προλαλήσαντες, ε, φαίνεται στην έκθεση πόσο καλή ή πόσο κακή είμαστε στον έλεγχο. Είχε μιλήσει ο κ. Μάρτιν Σούλτς ε, για το ότι στην Ευρώπη όλα κατά κάποιον τρόπο αποφασίζονται σε επίπεδο κορυφής. Ξέρετε τι σημαίνει όμως αυτό, ότι δεν υπάρχει διαφάνεια. Εμείς θέλουμε να εφαρμόζεται να εφαρμόζονται αυτά που λέει η συνθήκη της Λισαβόνας. Να είναι ανοιχτές οι συνεδριάσεις του Συμβουλίου. Να βλέπουμε και εκεί πώς κινείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και αυτό είναι κάτι όπου μπορούμε πράγματι να βελτιωθούμε. Να πούμε με απόλυτη σαφήνεια ότι και το Κοινοβούλιο μπορεί να καταστεί περισσότερο δημοκρατικό. Και να το πω αυτό, αυτό σημαίνει κατά κύριο λόγο ότι η δημοκρατία θα πρέπει να ισχύει ε, κατά την, ε, τον ορισμό των υποψηφίων που δεν υπάρχει σήμερα. Και κατά την άποψή μου εκεί ε, θα μπορούσαμε πράγματι να επιτύχουμε σημαντική βελτίωση. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. I don't Ευχαριστώ. Δεν έχω άλλους συναδελφούς που ζητούν το λόγο. Mercedes. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που αντικατέστησαν άλλους κοιόδες που δεν βρίσκονταν εδώ για να μπορέσουμε να συζητήσουμε την έκθεση. Οι παρατηρήσεις σας ήταν ενδιαφέρουσες. Οπωσδήποτε ένα από τα προβλήματά μας, τα βασικά μας προβλήματα και που θα μπορούσε να επιληθεί με μια διαθεσμική συμφωνία, αλλά απαιτεί όπως πολλά πράγματα και όπως θύμισε ο συνάδελφος Σέφλιν, ε, απαιτεί αλλαγές στις συνθήκες. Δυνατότητα πρόταση μορφή για έναν και μόνο επίτροπο ενδεχομένω ένα όπλο πυρηνικό που ε, εντάξει ως ε, πυρηνικό μόνο δεν θα χρησιμοποιηθεί αλλά χρειάζεται να δούμε την περίπτωση ε, μεταρρύθμισης αλλαγής στις, στις συνθήκες. Αυτό μπορεί να προταθεί στην έκθεση για να είναι και συνεπέστερη με όσες απόψεις εκφράστηκαν εδώ και να έχουμε και ένα ευρωστότερο θεσμικό σύστημα. Η ανανέωση στις συνθήκες, η αλλαγή στι συνθήκε, δεν χρειάζεται να περιπλέξει περαιτέρω τα πράγματα όπως έγινε με την όλη συζήτηση για τη Λισαβόνα και που ο σύστημα ε, περιέπλεξε την δουλειά μας σε πολλού τομεί, παρόλο που μας έδωσε περισσότερε αρμοδιότητες. Για το Συμβούλιο των Υπουργών τώρα, αυτό που είπε ο Ρίτσαρτ, είναι κάτι παραπάνω. Δεν είναι απλώς ε, πρόβλημα ορολογίας. Απλώς, αν το παρατηρήσετε προσεκτικά, οι υπουργοί που είναι μέρος του Συμβουλίου των Υπουργών είναι και εκτελεστές σε εθνικό επίπεδο των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα υπάρχει κάποιο είδους οριζόντιου ελέγχου, οριζόντιας επόψης για το πώ συγκεντρώνονται εκτελεστικέ αρμοδιότητε στα χέρια τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει βέβαια και το γεγονό ότι ε, από πάνω προς τα κάτω με του ίδιου υπουργού που εκπροσωπούν την εκτελεστική ε, εξουσία της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης, δηλαδή κάτι σαν την γερουσία, τη σύγκλιτο, ε, είναι αυτοί που θα φροντίσουν και για την εκτέλεση, την υλοποίηση της πολιτικής. Αυτοί κοιτάνε πώς εφαρμόζονται και όταν μιλάμε για κανονισμούς, αφού εγκριθούν οι οδηγίες, είναι εκείνοι που ακριβώς τις ε, εκτελούν, φροντίζουν για την εφαρμογή τους. Το πρόβλημα λοιπόν του ελέγχου, ε, του εγκάρσου, από πάνω προς τα κάτω ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα από τα προβλήματά μας ακριβώς γιατί ο έλεγχος από τι Εθνικές Βουλές δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στη λογική ελέγχου της ορθότητας της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου. Απέναντίας πολλέ φορές γίνεται με τρόπο αρκετά αμφιλεγόμενο σε σχέση με τα όσα ζητάει η Ένωση. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρόβλημα οποιοδήποτε ομοσπονδιακού ή παραμοσπονδιακού συστήματο, παραμένει όμω εξαιρετικά περίπλοκο σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, ακριβώ γιατί πολύπλοκη είναι και η φύση τη και αυτή των θεσμικών οργάνων. Βεβαίω, το πρόβλημα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι από αυτά που και σε επίπεδο πρακτικό και σε θεωρητικό όταν αρχίσουμε να συζητάμε την ενδεχόμενη αλλαγή στις συνθήκες, εκεί θα πρέπει να παρέμβουμε διότι το να οδεύει όλο ένα και περισσότερο στη λήψη αποφάσεων σε επίπεδο κορυφής η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως το είπε και ο κύριος Βίλαντ, είναι σαφώς ένα από τα προβλήματα. Από τα προβλήματα που μεταξύ άλλων αναδεικνύει με γλαφυρότητα την δυσκολία, την αδυναμία να ληφθούν αποφάσεις στην Ένωση. Διότι τελικά το Συμβούλιο προσπαθεί να λάβει αποφάσεις, συνεχίζει όμως να μεταφράσει σε πράξη, να δώσει σάρκα και οστά στις αποφάσεις που έχει λάβει. Αυτό είναι κάτι λοιπόν που θα πρέπει να επεξεργαστούμε. Βεβαίως, επίση ισχύει ότι ακόμη και αν έχουμε αρμοδιότητες περιορισμένες, αρμοδιότητες περιορισμένε για τον έλεγχο και την ε, επιβολή ποινών κυρώσεων, την τιμωρητική μας δηλαδή ε, λειτουργία, το Κοινοβούλιο έχει αναπτύξει πολύ τις ε, αρμοδιότητες να καθορίζουμε κάποια κατεύθυνση. Διότι ε, τουλάχιστον μπορούμε να καταδείξουμε κάποιες κατευθύνσεις ε, και ας μην έχουμε το, την αρμοδιότητα, το δίκαιο της πρωτοβουλίας. Και αυτό περιλαμβάνει κάποιες πραγματικές αρμοδιότητες. Εάν κοιτάξετε και μελετήσετε τις εθνικές βουλές, ποια είναι η σχέση τους με την εκτελεστική εξουσία, πολλές φορές τα εθνικά κοινοβούλια είναι πολύ πιο αυταρχικά. Δηλαδή, ε, όλο και περισσότερη εκτελεστική εξουσία έρχεται και παρεμβαίνει στη, στο πεδίο αρμοδιοτήτων των κοινοβουλίων, πολύ περισσότερο από ότι εδώ. Εάν κοιτάξουμε τα κείμενα των οδηγιών, τα νομοθετικά κείμενα που προκύπτουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και καταλήξουμε, μελετήσουμε τα τελικά συμπεράσματα. Βλέπουμε ότι είναι πολύ ισχυρό ο ρόλο του Κοινοβουλίου. Τα τελικά κείμενα πολύ συχνά είναι αρκετά τροποποιημένα χάρη στην παρέμβησή μα, κάτι που συμβαίνει πολύ λιγότερο στι εθνικέ βουλέ. Εκεί η βαρύτητα τη εκτελεστική εξουσία, τη πλειοψηφία ουσιαστικά εμ, απαλωτριώνει την ε, δυνατότητα δημοκρατικής ε, παρέμβασης των ε, υπόλοιπων βουλευτών της Εθνικής Βουλής. Άρα, νομίζω ότι εάν βοηθήσετε κι εσείς, στην έκθεση αυτή μπορούμε να υποδείξουμε τις κύριες γραμμές όπου χρειάζονται βελτιώσεις, όπου χρειάζονται ε, παρεμβάσεις, ώστε η λειτουργία μας αυτή να είναι λειτουργία ελέγχου της εκτελεστικής εξουσίας και διαφανέστερη ενώπιον των πολιτών μας και των εθνικών μας βουλών. Ίσως αυτό θα είναι μία από τις ε, βασικές μας ε, μέρημνες. Έχουμε πολλές προκλήσεις. Insieme al rapporto del collega Υπάρχει και το πρόβλημα των οργανισμών, δεν μπήκα σε λεπτομέρειες, διότι έχουμε και άλλη έκθεση εδώ, αλλά είναι σημαντικό να ρηλοσυμπληρωθούν οι δύο εκθέσεις και θεωρώ ότι εάν εργαστούμε παραλληλό και ε, για τις δύο, θα είναι ακριβέστατη και εξαντλητική η ανάλυση μας ω προ το ρόλο του Κοινοβουλίου και ως, ε, στη διάσταση του τιμωρητικού ελέγχου, του ελέγχου παρέμβαση και επιβολή κυρώσεων και τη του συμμαζέματο των εκτελεστικών εξουσιών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Να σας πω ότι 28 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα ε, έχουμε καθορίσει την εκπνοή της κατάθεσης, προθεσμίας κατάθεσης τροπολογιών και γύρω στα μέσα Ιανουαρίου θα γίνει η ψηφοφορία και μετά στην Ολομέλεια. 28 Νοεμβρίου 5 το απόγευμα. Και τώρα έχουμε τον κύριο Μέσελψη μαζί μας, άρα να ξαναπάμε στο σημείο 1 και να μας παρουσιάσετε την έκθεσή σας. Thank you so much. Um, Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους και τη γραμματεία για την ευελιξία που έδειξαν έτσι ώστε να γίνει η παρουσίαση του θέματος. Ξέρετε ότι έγιναν τρεις συστάσεις για την τροποποίηση του πρωτοκόλου 3. Η πρώτη είναι να μεταφερθεί στην, σε, στις διαδικασίες ε, ε, παρα πομπής ε, περί παραβιάσεων ε, και ε, μετά μια άλλη δυνατότητα έτσι ώστε να υπάρχει ταύτιση με τις αποφάσεις και μετά εναρμόνιση των ορισμών. Οι δύο πρώτες συστάσεις θα πρέπει να ακολουθηθούν γιατί δεν μπορούν δεν μπορεί κανείς να αντιτεχθεί σε αυτές, αλλά εάν μιλάμε για προσφυγή ε, σε καθαρά διοικητικές πράξεις, αυτό νομίζω ότι αποτελεί ε, αποτελεί παράβαση του συστήματος ε, που έχουμε πάντα, δηλαδή πρώτα ένα, ολοκληρώνεται ένα δικαστήριο και μετά μπορεί κανείς να προσφύγει σε άλλο δικαστήριο. Δεν πρέπει να παρεμβάλλονται οι διαδικασίες, προτείνω λοιπόν, να απορρίψουμε αυτό το τμήμα της πρότασης ε, έτσι όπως ακριβώς το λέω στην τροπολογία μου υπαριθμών 2. Το σημαντικό είναι να υπάρχει δυνατότητα να δείξουμε ανοιχτή διαδικασία. Το Κοινοβούλιο προχωράει γρήγορα, το, η Κομισιόν όχι τόσο πολύ. Ε, στην ουσία η Κομισιόν ε, έχει, ε, έχει πρόβλημα όσον αφορά την ανοιχτή διαδικασία και επομένως πολλές φορές επανειλημμένα και σίγουρα και με δική μου πρωτοβουλία έχουμε συζητήσει την Prudencia ε, και το απόρριτο του δικαστηρίου κυρίως ε, τα όσα, σε σχέση με τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 36 και από τα εθνικά δικαστήρια και από το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ε, είναι λογικό οι δικαστές να μην συμφωνούν σε ορισμένες περιπτώσεις ε, και ε, οι δικαστές της μειοψηφίας έχουν την δυνατότητα να εξηγήσουν τη θέση τους ε, με τον τρόπο αυτό που σαφηνίζεται ο νόμος κατά την άποψή μου. Και επομένως έχουμε καλύτερη νομολογία. Τα έχουμε ξανασυζητήσει στην Επιτροπή μας εδώ και υπήρξε συνένεση ε, ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσουμε για τη διαφάνεια ε, και την ε, ανοιχτή διαδικασία και μάλιστα ο εισηγητής Βίλκεν από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες από την Γιούρη. Ξέρω ότι συμφωνεί με την γενικότερη αυτή προσέγγιση. Και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να αναφερθεί και αυτό ε, και εδώ, έστω και αν ε, στη δικιά μου γνωμοδότηση θα πρέπει να ε, εξακολουθήσουμε να ασκούμε πίεση προς το δικαστήριο, μια και είναι το μόνο το μόνο θεσμικό όργανο το οποίο δεν έχει αυτό το άνοιγμα το οποίο προβλέπανε οι συνθήκες και αυτό νομίζω στο σύγχρονο κόσμο δεν είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτό. Χρειάζεται ε, ίδια, ε, ίδιος βαθμός ε, διαφάνειας όπως χρειάζεται και στα άλλα θεσμικά όργανα. Αυτά είχα να σας πω. Μπορούμε να προχωρήσουμε την επόμενη εβδομάδα γιατί από ό,τι καταλαβαίνω θα γίνει και ψηφοφορία την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε. Αλλά μια και έχουμε πολύ καλό πρώτερο βίο και είμαστε και γρήγοροι θα τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ πολύ. Για το ΕΛΚ υπάρχει κάποιος Σίλβια, θέλεις να μιλήσεις για τους σοσιαλιστές, έχω εδώ το όνομά σου. Θα ήθελα να ευχαριστώ θερμά τον συγητή μας. Ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να συζητηθούν κάποιες ε, τροπολογίες ε, κυρίως με τους συγητές. Αν τον κατάλαβα καλά, ε, δεν είναι ιδιαίτερα ενθουσιασμένος ε, σχετικά με το ερώτημα ότι οι αποκλίνουσες απόψεις θα πρέπει να δημοσιοποιούνται από την έκθεση. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει μια τελείως διαφορετική παράδοση και αυτό που βρίσκω καλό στις ε, προτάσεις του συναδέλφου Μέστερ Σμιτ είναι το θέμα ότι ε, πρέπει κανείς ε, να δει ε, πώς είναι δυνατόν στο μέλλον να επιτυγχάνεται καλύτερη εκπροσώπηση και των δύο φίλων στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ λίγες γυναίκες στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και εγώ στηρίζω την ιδέα να βελτιωθεί η κατάσταση όσον αφορά τα δύο φύλλα. Δεν ξέρω αν θέλετε εσείς να τοποθετηθείτε. Ε, δεν υπάρχει κανείς άλλος που να θέλει να λάβει το λόγο. Ως εκ τούτου, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Αν κανείς δεν λαμβάνει το λόγο, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει και καμία ε, αντίδραση. Θέλω να σας πω ότι την ε, καριέρα μου την πέρασα κατά το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα κάνοντας ακριβώς αυτό. Ανεξάρτητα από το πώς πρέπει να είναι η διατύπωση ή οτιδήποτε άλλο, νομίζω μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι ότι το να είναι κανείς ε, ανοιχτός, αυτό είναι κάτι ε, που πρέπει να υπάρχει στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως, είναι το δικαίωμα να υπάρχει αποκλίνουσα άποψη. Είναι δικαίωμα των πολιτών. Ε, στο Bundesverfassungsgericht στη Γερμανία, στο ανώτατο συνταγματικό δικαστήριο, όποιος αισθάνεται ότι πρέπει να εκφράσει μία διαφορετική άποψη, να μπορεί να το κάνει. Βεβαίω και προηγείται η άποψη του δικαστηρίου, αλλά μπορεί κανείς να εκφράσει τη διαφορετική του άποψη. Και πρέπει να πούμε ότι μερικέ φορέ ε, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ε, στι αποφάσει του, δεν υπάρχει σαφήνεια. Και γι' αυτό το λόγο σκεφτήκαμε να επιφέρουμε αυτές τις αλλαγές ε, στο πρωτόκολλο υπαριθμών 3. Κατά τη δική μου άποψη, αυτό που είναι σκόπιμο είναι να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια η ε, σαφήνεια μέσω της διαφάνειας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα θετικά που είπατε για τις άλλες τροπολογίες και θέλω να πιστεύω ότι ε, θα μπορούμε μετά από επικοδομητική συζήτηση να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Που λέει Πρόεδρος ε, θα είναι στις 29 Νοεμβρίου στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Μπάρμπαρα ε, που είναι η εφαρμογή των ε, δικαιωμάτων, ε, των συνταγματικών δικαιωμάτων. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχαν στην ερευνητική φάση Πιστεύω ότι αυτή, αυτός ο χάρτης, έστω και αν είναι νομικό, νομική υποχρέωση, εφαρμόζεται μερικώς και οπωσδήποτε έχει πολλές δυνατότητες που δεν τις έχουμε ακόμα διερευνήσει. Βεβαίως ξεκινάει η διαδικασία ε, από την ε, από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Παρ' όλα αυτά, κατά την άποψή μου, παραμένουν ακόμα φαίες ζώνες και επ' αυτών έχω ε, επικεντρωθεί. Να σας δώσω ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα. Είναι παράδοξο που ακόμα σήμερα σε πολλά νομοθετικά κείμενα πολύ σημαντικά η ενσωμάτωση έστω και μιας απλής αναφοράς του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων θα πρέπει να γίνει μέσα από τροπολογίες και δύσκολες διαπραγματεύσεις και η συμπερίληψη δεν φαίνεται ούτε δεδομένη ούτε ωφέλιμη από την αρχή της συγγραφής ε, του κειμένου. Πέρα από τους τυπικούς ε, περιορισμούς, βεβαίως το κείμενο δεν μπορεί να αποτελέσει την διεξοδικότερη των ε, ε, ερευνών ή ε, αναφορών, έστω και αν ε, ο χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων έχει πολύ συγκεκριμένο χαρακτήρα. Εγώ ε, έχω χωρίσει την παρουσίασή μου σε πέντε στοιχεία. Πρώτα απ' όλα η νομοθετική διαδικασία του, της Ευρωπαϊκής Ένωσης μια και ε, βάσει του άρθρου 51 της, ε, του, χάρτη αυτό αναφέρεται. Μέσω των μελετών προκύπτει ότι υπάρχει παθητική στάση απέναντι στην, ε, ε στον χάρτη και που δεν αφορά στην ουσία ούτε την πλήρη της εφαρμογή ούτε και την πρόθεσή της. Για το λόγο αυτό εγώ πρότεινα την δημιουργία άλλων νέων μηχανισμών που θα ευθυγραμμίσουν το ευρωπαϊκό δίκαιο με τις εξελίξεις του ε, δικαίου, του διεθνούς δικαίου και στις εκτιμήσεις αντικτύπου ε, να αναφέρεται με συγκεκριμένη αναφορά για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επίσης ε, λέω ότι θα πρέπει πέρα από τη διαδικασία δυνατότητα λήψη απόφασης θα πρέπει να υπάρχει παράλληλα ε, και ε, η διαρκής συμβολή ανεξάρτητων εξωτερικών ερευνών ε, και μελετών. Δεύτερον, οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ιδιαίτερη εστίαση στην εξωτερική δράση και την οικονομική διακυβέρνηση. Πρόκειται για θέματα τα οποία μπορεί να έχουν μεγάλη εμβέλεια και μπορούν ε, να ε, αναφέρονται σε πολλά ανθρώπινα δικαιώματα ε, με αποτελέσματα και αντίκτυπο εσωτερικό και εξωτερικό σε σχέση με τις τρίτες χώρες και σύμφωνα και με τις συστάσεις που ήδη έχουν κάνει άλλες, άλλα όργανα λέω, αναφέρω ότι θα πρέπει να υπάρξουν επιπλέον εχέγγυα ότι οι δικές εκτιμήσεις αντικτύπου για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να γίνονται πριν από την ολοκλήρωση των συμφωνιών. Η οικονομική διακυβέρνηση επίσης, λόγω των ιδιαιτέρων νοημάτων της, θα πρέπει να μελετηθεί ε, χωριστά. Ε, δηλαδή, στα συγκεκριμένα νομοθετικά ευρωπαϊκά εργαλεία ε, είναι σαφής. Επιπλέον ε, στοιχεία ε, και εργαλεία τα οποία θα πρέπει να προσθεθούν στα ήδη υπάρχοντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κεντρική θέση που ομάδες όπως το Eurogroup ας πούμε που δεν ελέγχονται από κανέναν δεν είναι δυνατόν να συνεχίζονται με τον τρόπο αυτό με ε, ε, διάφορους λοιπόν τρόπους, μερικούς από τους οποίους ανέφερα ήδη, ε, δεν έχει ενσωματωθεί ο χάρτης της νομοθετικής διαδικασίας. Ο Επίτροπος Ντούνα Μιάτοβιτς, υπεύθυνο για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στην έκθεσή του για την Ελλάδα ανέφερε ακριβώς την, την, ε, το μεγάλο πρόβλημα που η έλλειψη υποχρεώσεων ε, όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, μπορεί να δημιουργήσει σε κοινωνικά δικαιώματα και κυρίως το δικαίωμα για την υγεία. Όπως είπα και προηγουμένως, δεν υπάρχει δυνατότητα, δεν δεν υπάρχει ε, η υποχρέωση ε, αναφοράς ε, των κρατών μελών στον ε, χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων, πράγμα που οδηγεί σε δυνατότητα τα κράτη να μην εφαρμόζουν τον χάρτη. Και μάλιστα πολλοί είναι οι οργανισμοί οι οποίοι δεν ακολουθούν τις σωστές πρακτικές. Η πρότασή μας είναι να δημιουργηθούν οι βέλτιστες, ένας κατάλογος βελτίστων πρακτικών που θα πρέπει να, τους, να τις παρακολουθούν και να τις εφαρμόζουν όλοι οι οργανισμοί. Έστω και αν ε, ε, θεωρητικώς ε, τα κράτη συμφωνούν με, την, με τον χάρτη και έστω και αν δεν τον έχουν προσυπογράψει όμως, παρόλα αυτά δεσμεύονται από τα όσα στο χάρτη αναφέρονται. Κατά την έννοια αυτή προσπαθούμε μέσω της εκθέσεως να υπερβούμε τις ελλείψεις που έχουμε διαπιστώσει όσον αφορά την γνώση για τον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων, προτείνοντας συγκεκριμένα μέτρα ε, τα οποία θα βοηθήσουν τα κράτη-μέλη στην υλοποίηση του χάρτη. Επόμενο σημείο, η εμβέλεια, το πεδίο εφαρμογής του χάρτη. Η ερευνητική δραστηριότητα κατέδειξε τις δυσκολίες κατανόησης ή πλήρους κατανόησης στον τρόπο λειτουργίας του άρθρου 51 ε, του χάρτη και όσον αφορά την ε, ε την διχοτόμηση από τη μία καθήκον αποχής από την άλλη καθήκον λήψης μέτρων που δεν αναφέρεται σε άλλα ανάλογα εργαλεία διεθνούς δικαιώματος αλλά και όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής ε, του χάρτη ε, από τα κράτη-μέλη. Είναι δυσκολίες ε, οι οποίες έχουν αντίκτυπο και στην δυνατότητα προώθησης με ομοιόμορφο τρόπο των δικαιωμάτων που αναφέρονται ήδη στο χάρτη, αλλά και όσον αφορά την συγκεκριμένη χρήση του χάρτη από τους ε, σε εθνικό επίπεδο και από τους ε, εμπλεκόμενους. Επομένως θα πρέπει να υπάρξει μια κοινή προσπάθεια έτσι ώστε ε, να γίνει γνωστός ο χάρτης έτσι ώστε να καταφέρουμε μία μέρα κάποια στιγμή να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε αλλά και να υπερβούμε τα όσα στο άρθρο 51 αναφέρονται. Ευχαριστώ πολύ όλους ε, και ευχαριστώ εκ των προτέρων για τα σχόλια, αν και βλέπω ότι απουσιάζουν οι shadows, οι σκιώδεις. right? Yes. Αμέσως να σας ρωτήσω αν θέλετε να μιλήσετε. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και την Μπάρμπαρα. Ευχαριστώ για την δουλειά σου. Είναι ένα θέμα που μας ενδιαφέρει στην Επιτροπή εδώ και αρκετό καιρό. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό εδώ στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων και πριν τις ευρωεκλογέ να καταφέρουμε να υποβάλουμε μια ποιοτική έκθεση. Είναι η ίδια η χάρτα το αντικείμενο της έκθεσής μας. Η χάρτα είναι το κατεξοχήν έγγραφο ε, το πλέον σημαντικό έγγραφο που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Αυτό καθορίζει τα δικαιώματα των πολιτών. Αφορά αυτού του ίδιου του πολίτε. Και όχι απλώ τα δικαιώματά του, αλλά τα δικαιώματα κάθε ανθρωπίνου όντω, ανδρών και γυναικών που ζουν στην επικράτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η ουσία τη ευρωπαϊκή ε, διάσταση και ε, ω προ του πολίτε ακριβώ, ε, το Κοινοβούλιο πρέπει να παρακολουθεί, να επαγρυπνεί ώστε η καρδιά της Ευρώπης να χτυπά με καλό ρυθμό. Ε, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενσαρκώνουν ακριβώς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει λοιπόν να σέβονται πλήρως τις διατάξεις της χάρτας και θα πρέπει να εφαρμόζουν όλες τις αρχές της. Θα συμφωνήσω απολύτως με την εισηγήτρια. Η υλοποίηση από τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Χάρτα και των διατάξεων τη, έχει πάρει καλή κατεύθυνση. Το λέει και στην έκθεσή τη και συμφωνώ. Είναι σημαντικό τα θεμελιώδη δικαιώματα να ενισχυθούν. Και ο οργανισμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων σίγουρα διαθέτει ε, ειδικέ γνώσεις, τις οποίες θα μπορούσαμε να αξιοποιούμε καλύτερα. Και δύο σημεία τα οποία μου είναι ιδιαίτερα προσφυλή και για τα οποία θα προτείνω οπωσδήποτε τροπολογίες. Πρώτον το σημείο 6. Η εισηγήτριά μας επιθυμεί συστηματική εξπόστ αξιολόγηση και εξακρίβωση του κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί την ε, συμβατότητα των διατάξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις διατάξεις της Χάρτας των Θεμελιωτών Δικαιωμάτων. Υπάρχει ρήτρα αναθεώρησης ε, για την ε, χάρτα που δεν περιλαμβάνεται σε όλα τα νομοθετικά κείμενα. Πρέπει να πω ότι δεν είμαι εγώ εισηγητρία βεβαίω, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι αυτή η προσέγγιση που πρέπει να επιλέξουμε. Δεν μπορούμε απλώς να επιλέξουμε αυτήν την προσέγγιση, διότι έρχεται να δημιουργήσει αντίφαση με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Οι νομοθέτες που θα έχουν παραβιάσει την ε, νομοθεσία όπως προκύπτει από την χάρτα θα πρέπει να ε, κρίνονται βάσει μια συγκεκριμένη διαδικασία και μετά η υλοποίηση θα μπορούσε να διορθωθεί στο μέσο της διαδικασίας. Δεν νομίζω ότι είναι σωστά συντεταγμένο το σημείο 6. Κάθε κράτος θα πρέπει να καθορίζει τη δική του νομοθετική πορεία και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παρακολουθούν το σεβασμό των διτάξεων της χάρτας. Αυτό είναι αυτονόητο. Απλώς πρέπει, νομίζω, να μην υιοθετείται καν μια νομοθετική πράξη εφόσον ε, αντιφάσκει με τα όσα προβλέπει η χάρτα. Το 16 τώρα για του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εκεί Καλό θα ήταν λίγο να το ξαναδούμε. Ε, νομίζω ότι η συγγήτριά μας υπερβάλλει λίγο προς το ρόλο των οργανισμών. Στο σημείο 16 λέγεται ότι οι οργανισμοί έχουν πολύ σημαντικές δυνατότητες που θα τους επιτρέψουν, θα επιτρέψουν μάλλον στα κάτι μελη να παρακολουθούν τις υποχρεώσεις που εκπηγάζουν από τη χάρτα. Αυτό όμως το τεράστιο δυναμικό των οργανισμών Από πού προέρχεται, θα καταργήσουμε τους δορυφορικούς οργανισμούς, θα καταργήσουμε τον οργανισμό των σιδηροδρόμων. Ε, Θα πρέπει να δούμε εάν παρακολουθείτε σωστά η συμμόρφωση με τις διατάξεις της χάρτας. Άρθρο 51. Και εδώ βλέπω να υπάρχει ανάγκη για συζήτηση και προφανώς ε, και προφανώς ε, ε, πρέπει να δούμε όλα αυτά τα άρθρα. Έχω την εντύπωση ότι το άρθρο 51 πολύ συχνά παρερμηνεύεται ή για να το πω ε, διαφορετικά, ότι ερμηνεύεται διαφορετικά. Ε, αν δει λοιπόν κανείς το κείμενο και την ε, επεξήγηση του χάρτη βλέπει ότι το άρθρο 51 κατ' ουσίαν το μόνο που κάνει είναι να ορίζει το πεδίο εφαρμογή του χάρτη. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, τις αρμοδιότητες που ορίζονται από τις συνθήκες, η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έχει αρμοδιότητες που τις έχουν μεταβιβαστεί από τα κράτη-μέλη και αυτό αναφέρεται με απόλυτη σαφήνεια στο κείμενο. Ο χάρτης αυτός πέρα από τις μεταβιβαστήσεις αρμοδιότητες δεν προβλέπει άλλες αρμοδιότητες για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, τα θεμελιώδη δικαιώματα όπως είναι παγιωμένα και αναφέρονται στο χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ε, με ε, τη συμφωνία αυτή καθίστανται ενεργά. Βεβαίως εκεί μπορεί κανείς ε, να βάλει ένα ερωτηματικό, αλλά κατά την άποψή μου αυτό δεν αλλάζει τίποτα στο γεγονός ότι ο χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων δεν είναι χάρτης για τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη έχουν όλα τις δικές τους, τους δικούς τους κανονισμούς περί δικαιωμάτων. Και κάτι άλλο. Στο κείμενο γίνεται λόγος για το ότι όσον αφορά τον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων ε, πρέπει να υπάρξει ε, μία προσπάθεια για καλύτερη νομοθέτηση, better law making. Εγώ δεν ξέρω τι πιστεύουν οι άλλες πολιτικές ομάδες, αλλά εγώ πιστεύω ότι αυτή η νέα ρύθμιση αποφασίστηκε σε αυτή την νομοθετική περίοδο με μεγάλη πλειοψηφία και νομίζω ότι ε, θα ήταν πάρα πολύ δυσάριστο αν δεχόμασταν ότι κάναμε κακή δουλειά και ότι πρέπει να επαναδεπραγματευτούμε όλη αυτή τη συμφωνία. Εγώ λοιπόν σε αυτό το θέμα δεν συμφωνώ. Παρόλα αυτά, παρά την κριτική που μόλις τώρα άσκησα, θα ήθελα ειλικρινά να ευχαριστήσω πολύ θερμά για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε, ε, για πολύ καλές ε, προτάσεις ε, και προσβλέπω στην συνέχιση της καλής συνεργασίας έτσι ώστε την έκθεση αυτή να την προχωρήσουμε ικανοποιητικά μέχρι το τέλος της θητείας μας. Ευχαριστούμε Σιλβί, δεν βλέπω άλλους κοιόδης εδώ. Δεν βλέπω κανένας να θέλει να μιλήσει εκ μέρους όσων λείπουν. Μπάρμπαρα, Πολύ σύντομα να ευχαριστήσω θερμά τη Σιλβή για αυτά που είπε και για τις προτάσεις της. Φυσικά δεν συμφωνώ με όλα. Αλλά θεωρώ ότι μέσα από διάλογο Θα δούμε αν υπάρχουν κάποια σημεία σύγκληση, ιδίω για του οργανισμού. Ίσως μπορούμε να δούμε ποιοι οργανισμοί έχουν τέτοιο ρόλο στον τονισμό των εθνικών πολιτικών. Γιατί όπως λέτε, Σιλβί, σωστά, μερικά, μερικοί δεν έχουν κανένα τέτοιο ρόλο. Ως προς το άρθρο 51 το 51. Περιμένω να δω τις σχετικές τροπολογίες. Φαντάζομαι ότι θα είναι τροπολογία ε, διαγραφής της δυνατότητας. Αναθεώρησης της συνθήκης. Εγώ θεωρώ ότι μπορεί να πάει κανείς πέρα από το άρθρο 51. Αλλά αυτό θα το συζητήσουμε. Μια συντομότατη παρατήρηση για αυτό που είπε η Σιλβή. Και είναι απλώς ένα παράδειγμα για τις διαθεσμικές συμφωνίες, αλλά δεν είπα σε καμία περίπτωση ότι η δουλειά έχει γίνει στραβά. Ξέρω ότι η δουλειά έχει προηγηθεί για το δοσχέ αυτό. Δεν πιστεύω λοιπόν ότι έχει γίνει κακή δουλειά. Απλώς πιστεύω ότι επειδή ο κόσμος αλλάζει, τα προβλήματα πολλαπλασιάζονται, η ιστορία προχωρεί, ίσως λοιπόν θα μπορούσαμε να σκεφτούμε και βελτιώσεις της καλής δουλειάς που ήδη έχει γίνει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Στη φάση αυτή κλείνουμε τη συζήτηση για το θέμα. Α, θέλετε να πείτε κάτι ακόμα. Έχουμε χρόνο, βεβαίω. Μία ερώτηση έχω μόνο να κάνω. Μπορείτε να μας πείτε και την καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση τροπολογιών. Θα μπορούσα να το κάνει, αλλά θα το κάνω εγώ. Προθεσμία 3 Δεκεμβρίου, στις 5 το απόγευμα. 3 Δεκεμβρίου, 5 το απόγευμα, σε δύο περίπου εβδομάδες νομίζω, έτσι. Αυτό που πρέπει να αποφασίσουμε τώρα είναι εάν μας κάνει αυτή η προθεσμία και μετά έχουμε και την συνεδρίαση του Γενάρη για να δούμε τις τροπολογίες αυτές, την ψηφοφορία στην ΑΦΚΟ το Φεβρουάριο. Αργά δεν είναι για ολομέλεια. Ελπίζω θα τα καταφέρουμε για το Μάρτιο. Υπάρχει χρόνος γι' αυτό, πολιτικός ελπίζω να είναι δυνατόν. Δεν υπάρχει λόγος να μην προλάβουμε. Αλλά δεν μπορώ να δώσω παράταση. Μερτσέντες. Νομίζω ο Μάρτιος δεν θα είναι κάτι το εφικτό. Θα τον έχουν ε, μπλοκάρει για νομοθετικές πράξεις. Το Φεβρουάριο πρέπει να περάσει αυτή η έκθεση πρωτοβουλίας. Δεν ξέρω αν είναι η λιμένη απόφαση, αλλά σίγουρα είναι κάτι που ισχύει τώρα. Θα ληφθεί. Δεν έχει αποφασιστεί κάτι ακόμα. Έχουμε όμως δύο ολομελίες το Μάρτιο. Θα το κοιτάξουμε. Διότι αν ισχύει, θα πρέπει να ξανασκεφτούμε το χρονοδιάγραμμα. Η προθεσμία για την υποβολή των απολογιών πάντως δεν αλλάζει. 3 Δεκεμβρίου, 5 το απόγευμα. Απλώς ίσως να έχουμε και καμιά έκτακτη συνεδρία, θα το δούμε. Right. Να το σκεφτούμε, διότι αν η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών μείνει 3 Δεκεμβρίου, μετά είναι 6 ε, του μήνα η εξέταση των τροπολογιών. Μήπω προτιμά να γίνει η εξέταση των τροπολογιών 6, Γενάρη, αντί για το 6 Δεκέμβρη αντί για το Γενάρη. Δεν θα έχουμε μεταφραστεί όλα. Θα είναι λίγο δύσκολο τώρα. Αλλά θα έχουμε περισσότερο χρόνο. Συνάδελφοι, θα διακόψω τη συνεδρίαση. Το Γενάρη θα ψηφίσουμε στην ΑΦΚΟ, οπότε θα περάσει στην Ολομέλεια το Φλεβάρι. Έχουμε δύο συνεδριάσεις το Γενάρη. Κάτι θα καταφέρουμε. Τώρα θέλω να διακόψω τη συνεδρίαση. Θα ψηφίσουμε στις 11. Δεν έχουμε τίποτα μεταξύ. Και δεν υπάρχει και κανείς στην αίθουσα. Τα λέμε στις 11.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

Αυτός είναι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

Θα ήθελα να ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες. Να σας ενημερώσω ότι ένα από τα σημεία ε, στον κατάλογο των ψηφοφοριών, η έκθεση του κ. Κόρμπετ, επειδή είχαμε ζητήσει από την νομική υπηρεσία να τοποθετηθεί και η γνωμοδότηση έφτασε μόλι στα χέρια μα και πολλοί συνάδελφοι δεν πρόλαβαν να διαβάσουν και υπάρχουν εκκρεμή ζητήματα και μπορεί να υποβληθούν και νέε τροπολογίε. Τα κοιτάμε λοιπόν και ίσω να γίνει και συνεδρία των σκιωδών αυτή την εβδομάδα. Οπότε προτείνω αναβολή τη ψηφοφορία για την επόμενη εβδομάδα. 27 του μήνα. 26, 26 να με συγχωρείτε. Α, Α, όχι, 6 Δεκεμβρίου. Δεν μπορείτε. Μπορείτε ή δεν μπορείτε. Ναι, ναι, μπορώ στις 6 Δεκεμβρίου. Α, εγώ νόμιζα το Νοέμβριο. Επειδή λοιπόν ο εισηγητή μα μπορεί να είναι παρόν μόνο στι 6 Δεκεμβρίου, θα ψηφίσουμε στι 6 Δεκεμβρίου. Can we accept that? Μπορείτε να το δεχτείτε. Ε, on this point. Για αυτό το σημείο. Max, yes, please. Max. I find it strange. Το βρίσκω περίεργο να αναβάλουμε αυτή την ψηφοφορία κατά αυτόν τον τρόπο. Η νομική υπηρεσία ε, έχει συντάξει τη γνωμοδότησή της εδώ και καιρό, ακόμα και αν δεν είχε δημοσιευτεί μέχρι χθε. Εγώ την έλαβα χθε και ο κόσμος θα έπρεπε να την είχε διαβάσει. Και να την αφομοιώσει Υπάρχει κίνδυνος. Οι θετικές επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει η ψηφοφορία μας στις υπόλοιπες διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην ε, γίνουν πραγματικότητα. Διότι θα χάσουμε τον αγώνα δρόμου της Αυστριακής Προεδρίας. Νομίζω πιο ε, σοφό θα ήταν και πιο αποτελεσματικό να ψηφίσουμε τώρα, αντί να αναβάλουμε. Ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Άλλος, Χέλμουτ. Uh, I would agree with what Ναι. Συμφωνώ με τον Μαξ, διότι έχουμε προετοιμαστεί πάρα πολύ προσεκτικά. Ε, και την γραμματοδότηση την λάβαμε χθε. Είχαμε χρόνο να την κοιτάξουμε. Άλλωστε, είχαμε προγραμματίσει την παρουσία μα εδώ. Εγώ στι 6 δεν θα βρίσκομαι εδώ, γιατί θα είμαι στη Γενέβη σε συνεδρίαση του ΠΟΕ, σε κοινοβουλευτική συνέλευση. Οπότε η αναβολή θα δημιουργήσει πρόβλημα. Εγώ προτιμώ να ψηφίσουμε σήμερα. Άλλα σχόλια από αυτού. Yes, Mr. Wieland. Κύριε Βίλαντ. Εμείς υπέρ της αναβολής. You will have to say it once again. για τους λόγους που ανέφερε και η Πρόεδρος. Γι' αυτό εμείς θέλουμε να αναβληθεί η ψηφοφορία. Δεν κατάλαβα τι έγινε, αλλά κατάλαβα ότι προτείνατε την αναβολή. Υποστηρίζετε τη δική μου την πρόταση ως Πρόεδρου. Γιο Κοιτάξτε, όποιος βιάζεται σκοντάφτει. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να σας πω ότι μπορούσαμε να το διαβάσουμε το όλο θέμα μεμονωμένα, αλλά όχι ως ομάδα. Και λυπάμαι που δεν μπορούμε να ψηφίσουμε σήμερα. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όσον αφορά τον κανονισμό. Γι' αυτό ε, να αναβάλουμε στις, για τις 6 Δεκεμβρίου. Άρα και εσείς στηρίζετε την αναβολή, ε? Οπότε νομίζω ότι έχουμε πλειοψηφία υπέρ τη αναβολή. Ναι, ω εισηγητή, εγώ θα δεχτώ την απόφαση της Επιτροπής. Ε, υπομονούσα για τη σημερινή ψηφοφορία. Η γνωμοδότηση της Νομικής Επιτροπής θεωρεί μόνο μία τροπολογία αντίθετη με τον νόμο, αλλά αν αναβάλουμε, ας αναβάλουμε, να το αξιοποιήσουμε και θα κοιτάξω να συνεδριάσω με τους κοιόδης μου, μήπω βρούμε λύση για τις αναπομείνασες δυσκολίες. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Να αποφασίσουμε λοιπόν υπέρ της αναβολής. Και τώρα να κάνουμε ένα τεστ με τις κάρτες και τα μηχανήματα. The vote is, the test vote is open. Δοκιμαστική ψηφοφορία. So could you please check your capacity? We are 20, 20 21, 20.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 Ωραία, λοιπόν, αρχίσουμε τις προφορίες. Ξεκινάμε με το σχέδιο έκθεσης για τη διαφοροποιημένη παρέμβαση του κυρίου Ντιράν. Επίσης θέλουμε και σιωπή για τις προφορίες. 31. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Οίκον 1, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 4, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 37, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 38, υπέρ, κατά, έλεγχος για την 38, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας, Απορρίπτεται. 11 προς 11. Συμβαστική 5. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 42. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Έκον 6. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 43. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 44. Υπέρ, κατά, αποχές, ελέγχουμε για τη 44. 11 προς 11 απορρίπτεται. 6. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Budget 5 υπέρ κατά Δεν καταλαβαίνω. Για να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 11 προς 11 πάλι. Σήμερα έχουμε καλή πλειοψηφία. Έκον 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβεστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 74 ε, υπέρ, 74 υπέρ, κατά. Οι σοσιαλιστές είναι κατά. Να εξακριβώσουμε, να κάνουμε έλεγχο. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται 14 προς 8 75 υπέρ κατά να ελέγξουμε για την 75 πέρας απορρίπτεται 10 προς 12 78 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 76 υπέρ κατά έλεγχος για την 76 άρχεται η ψηφοφορία Δευτέρας. 11 προς 11 απορρίπτεται. 77 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται 9 προς, 10, προς 13. Προφορική τροπολογία 1. Είναι κανείς κατά. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 11. 10, συγγνώμη. Υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε για τη συμβαστική 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Δύο δεν θέλουν να ψηφίσουν από ό,τι φαίνεται, αλλά πρέπει να κλείσουμε την ψηφοφορία έτσι κι αλλιώς. Την κλείνουμε. 7 προς το 10 απορρίπτεται. 11, συμβαστική 11. Όχι. Α, ναι, 79. Υπέρ. Ψηφίζουμε αυτέ που περιλάμβαναν, περιλάμβανε η 79 υπέρ. Κατά. Έλεγχο για την 79. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 15 προ 7. Συνάδελφοι, έπρεπε να σα πω να ψηφίσουμε και την 80 και την 81 μαζί, γιατί είναι πανομοιότυπες ε, οι δύο ε, Οι υπόλοιπε εκπίπτουν, μου λέει η γραμματέας, ε, συμβαστική 11 υπέρ. Κατά, αποχέ. είμαστε διχασμένοι να ελέγξουμε για την 11. Πέρας. Απορρίπτεται 10 προς 12. 87 υπέρ κατά να ελέγξουμε για τον 87. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται 10 προς 12. 86. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 88. Υπέρ, κατά, έλεγχος για τον 88. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται 10 προς 10. 89 και 90 ταυτόσιμες υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 91 υπέρ. Όχι. Εκπίπτει. Καταπίπτει. 2 υπέρ. 2, 2. 2. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος για την 2. Πέρας. 10 προς 12 απορρίπτεται. Τροπολογία πρώτη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 4. Έλεγχος για την 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 10 προς 12. Συμβαστική πρώτη υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 8 υπέρ. Κατά. Έλεγχος για την 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 9 προς 13. 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά εποχέ εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά. Παρακαλώ. 14. Τι. Υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά. Έλεγχο για το 15. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται 11 προς 11. 16. Καταψήφισατε δικιά μου την τροπολογία. Την καταψηφίσατε. Λάθος. Μέα κούλπα. Μπορείτε απλώ να ζητήσετε από την γραμματεία να αλλάξει την ψήφο σα στα πρακτικά, αλλά δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα αποτέλεσμα τη ψηφοφορία. Μην κάνετε έτσι, Πασκάλ, και σε εσά έχει συμβεί. Μπορεί να καταγραφεί, αλλά δεν μπορούμε να ξαναψηφίσουμε. Δεν αλλάζει το αποτέλεσμα στην Ολομέλεια, κύριε Μπρόκ. Μετά από 14 χρόνια πρέπει να το ξέρετε. Sorry, Πάολο. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Πάμε στην 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. απορρίπεται. 17. Υπέρ. Έλεγχος για τη 17. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται 11 προς 11. Χέλμουτ, ελπίζω να μην καταψήψεις την ίδια στην τροπολογία. 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21 Παύλο, προσοχή. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ. Να ελέγξουμε για την 25. Άρχεται η ψηφοφορία. Α, δεν είχε ξεκινήσει. Τώρα ναι. Πέρασε. 11 προς 10 πέρασε. Εγκρίνεται. 26 υπέρ. Κατά αποχές. Έλεγχος για την 26. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Να απορρίπτεται. 10 προ 12. 26. 27 τώρα υπέρ. Κατά αποχέ. Απορρίπτεται. 28 υπέρ. Έλεγχο για την 28 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 12 προς 10. 29 υπέρ. Κατά αποχές. Έλεγχος για την 29. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται 8 προς 14. 30 υπέρ κατά αποχές. Ελέγχουμε για τα 30. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 9 προς 13. Όλες οι εναπομένες αστροπολογίες είναι εκτός θέματος. Τελική λοιπόν ψηφοφορία της έκθεσης όπως τροποποιήθηκε, ονομαστική ψηφοφορία. «20 προς 2 εγκρίνεται. Πάρα πολύ καλά. Συγχαρητήρια, κυρία Ντουράν. κύριε ε, συγχαρητήρια, Πασκάλ. Και τώρα η έκθεση του κυρίου Σόλτς για την προστασία του ε, ενωσιακού προπολογισμού σε περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων σε ό,τι αφορά το κράτο δικαίου ε, στα κρατή-μέλη. Ξεκινάμε με την 28. Τι έγινε. Για να ξεκινήσουμε. 28. Το κύριο Γκέγκολτ. Έκθεση Σόλτ. Η πρώτη τροπολογία είναι υπέρ 28. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 7A υπέρ κατά αποχές ε, να ελέγξουμε την 7α. Ε, ψηφίζουμε παρακαλώ. Επτά αλφα. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Δεν την έχουμε ακόμα κλείσει την ψηφοφορία. Ποιο είναι το πρόβλημα. Ψηφίσατε ήδη ε, στο 7α, έκλεισε η ψηφορία και απορρίφθηκε 11 προς 11, 65. Υπέρ Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Το 63 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε για την 63 που μοιάζει να εγκρίνεται. Η 63 παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία και απορρίπτεται. Ε, η 64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 11 υπέρ κατά ε, ελέγχουμε την 11 ψηφίζουμε παρακαλώ έκλεισε ψηφοφορία και απορρίπτεται 9 προς 12 η 66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 68 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 69 υπέρ υπέρ οι σοσιαλιστές ελέγχουμε την 69 ψηφίζουμε παρακαλώ έκλειση ψηφοφορία απορρίπτεται η 70 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται 71 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 72 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 73 υπέρ ελέγχουμε την 73 ψηφίζουμε παρακαλώ Έκλειση ψηφοφορία απορρίπτεται 9 προς 12. Και τώρα πάμε στην 74. Υπέρ κατά απορρίπτεται. Η 12 υπέρ κατά εγκρίνεται. Η 75 υπέρ κατά απορρίπτεται. Η 76 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 77 υπέρ κατά απορρίπτεται. 78 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, η 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, η 81 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, η 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 82 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, η 83 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, η 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 84 όχι, 85 υπέρ κατά ελέγχουμε την 85. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Πάμε στην 86. 87 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 88 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 89 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 90 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 93 υπέρ Η 93 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Η 98 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 99 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 19 υπέρ, όχι, η 11 καταπίπτει. Πάμε στην συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 101 για αυτήν ψηφίσαμε. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. στην 25 πάμε τώρα. Λοιπόν, πάμε στην 25 παρακαλώ. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 113. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η συμβιβαστική 13. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 118 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 116 και η 117 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 119 υπέρ κατά απορρίπτεται. Για την 120 ψηφίσαμε απορρίπτεται 120 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 121 υπέρ κατά ελέγχουμε για την 121 ηλεκτρονικά εγκρίθηκε η συμβαστική 1 Η 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, η 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, η 3 υπέρ κατά για την 3. Ελέγχουμε για την 3. Έκλεισε ψηφοφορία και απορρίφθηκε η 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, η 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, η 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, η 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, η 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, η 40 υπέρκατα αποχές απορρίπτεται, η 41 υπέρκατα αποχές απορρίπτεται, η 42 υπέρκατα αποχές απορρίπτεται, η 43 υπέρκατα αποχές εγκρίνεται, συμβαστική 2 υπέρκατα αποχές εγκρίνεται, η 44 υπέρκατα αποχές ε, απορρίπτεται, η 47 ηλεκτρονική επαλήθευση για τις 47. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε. Απορρίπτεται 11 προς 11 η 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η συμβαστική 4 υπέρ κατά εγκρίνεται. Η 5 η συμβαστική υπέρ κατά εγκρίνεται. Η 54 υπέρ κατά εγκρίνεται. Η 55 υπέρ κατά εγκρίνεται. Η 56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά εγκρίνεται. Η 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τελική ψηφοφορία ψηφίζουμε παρακαλώ έκλειση ψηφοφορία Περνάμε τώρα την γνωμοδότηση της κυρίας Ταπαρδέλ σχετικά με την φορολογική πιθανότητα Υπάρχει μία προφορική τροπολογία. Δεν είναι όμως εδώ. Επομένως δεν μπορεί να παρουσιάσει προφορική τροπολογία. To ε, θα τα πεις εσύ. επειδή δεν είναι παρούσα η προφορική τροπολογία είναι να απορριφθεί αυτή η έκθεση. Ε, you finished, αυτό ήθελες να πεις μόνο γιο. Θέλει να πει κάποιος ε, άλλος κάτι. Ναι, πρόταση λοιπόν να ε, απορριφθεί η πρόταση αυτή. Αυτή είναι η προφορική τροπολογία. Εγώ θα ήθελα εξ του ΕΛΚ να εκφράσω την αντίδρασή μου. επομένω ψηφίζουμε. Όχι, δεν ψηφίζουμε. Δεν ψηφίζετε την προφορική τροπολογία. Θέλετε να ψηφίσουμε την έκθεση. Πολύ ωραία. Θα ψηφίσουμε για την έκθεση κανονικά, λέει η Πρόεδρος. Τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται.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 πέρας της ψηφοφορίας και απορρίπτεται 10 υπέρ 11 κατά. Τροπολογία 11 υπέρ, κα, ε, υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται η επόμενη... Δεν ψηφίζεται όλοι ομόφωνα, επομένως... Πέρασε απορρίπτεται. Η τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές ε, ηλεκτρονική επαλήθευση. Έτσι εδώ φαίνεται τα πάνω κάτω. Η, το ΕΛΚ ψηφίζει τις τροπολογίες του, των σοσιαλιστών, οι σοσιαλιστές αντίστοιχα των ε, ε ΕΛΚ και τα λοιπά. Εν πάση περιπτώσει απορρίπτεται 11 υπέρ 11 κατά. Ε, πηγαίνουμε τώρα στην τροπολογία 3 απευθείας. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και απορρίπτεται 10 με 12. Ψηφίζουμε για την τροπολογία 4. Και εδώ δεν έχουμε ομοιόμορφη, ε, ομοιόμορφη τρόπο ψηφοφορίας, άρα ηλεκτρονική επαλήθευση. Πέρας απορρίπτεται. Τροπολογία 5, να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας, απορρίπτεται τελική ψηφοφορία όσον αφορά το σύνολο της γνωμοδότησης ε, διονομαστικής ε, κλίσεως. Άρχεται η ψηφοφορία. Μπορούμε να ολοκληρώσουμε. Εγκρίνεται. 11 με 10. Γιολάινεν. Εγκρίναμε την ε, έκθεση αυτή, αλλά ο Γιολάινεν θέλει να πάρει το λόγο. Η κυρία Ταπαρδέλα θα ήθελε να αφαιρεθεί το όνομά της από την έκθεση αυτή. Ναι, ναι, είναι τρέχουσα πρακτική. Το καταλαβαίνω. Θέλει κάποιος άλλος να το αναλάβει. Συνήθως, εθιμικά και τα λοιπά, ο πρόεδρος ε, αναλαμβάνει την έκθεση σε τέτοια περίπτωση, αλλά η πρόεδρος έχει την αντίστοιχη εγνωμοδότηση στην ΕΚΟΝ. Επομένως, ε, θέλει κάποιος εθελοντικά να βάλει το όνομά του. Ναι, ναι, εγώ, εγώ. Εκτός και αν κάποιος από του σοσιαλιστές θα ήθελε να πάρουν τη θέση αυτή. Ω, τι ευγενεί που είστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, χαίρομαι γιατί μου κάνετε ένα τόσο πρώιμο ε, δώρο χριστουγεννιάτικο. Τελευταία. Ζωζέπ Μαρία Τέρι Κάμπρας ε, σχετικά με τα προγράμματα Rights και Values. Ξεκινούμε. Τροπολογία 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 55 ε, θα κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση άρχεται η ψηφοφορία Ζωζέπ ψήφισε και εσύ πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται 3 ψήφοι υπέρ, 19 κατά. Τροπολογία 54 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 56 ε, και 57 ταυτόσημες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 5 ε, ηλεκτρονική επαλήθευση για το 5 άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 12 ε, υπέρ 10 κατά επόμενη τροπολογία θα είναι η 58 Α, ναι, γιατί η άλλη καταπίπτει. 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση επί της τροπολογίας 9 άρχεται η ψηφοφορία πέρας 11 ε, υπέρ 11 κατά απορρίπτεται 64 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται οι σοσιαλιστές ήταν υπέρ όχι α τότε να κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση επί της τροπολογίας 64 ε, άλλη μία ψήφο χρειάζομαι πρέπει άλλος ένας να ψηφίσει κάποιος ξέχασε 12 υπέρ 10 κατά εγκρίνεται Πάμε στην τροπολογία 10 υπέρ. Ε, να γίνει η ηλεκτρονική επαλήθευση επίσης επί του 10 γιατί δεν είναι ε, ομοιογενής η ψηφοφορία. Πέρας. 15 υπέρ, 7 κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 65 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 11 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ. Και εδώ θα πρέπει να γίνει ηλεκτρονική επαλήθευση. Δεν είναι ομοιογενής ο τρόπος ψηφοφορίας. Ψηφίστε όλοι ε, πέρα της ψηφοφορίας και απορρίπτεται 7 υπέρ 15 κατά. Τροπολογία 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 15 υπέρ ε, θα πρέπει να γίνει με ηλεκτρονική ε, ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 9 υπέρ 13 κατά. Τροπολογία 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 79 όχι, 79 καταπίπτει, περνάμε στην 90 υπέρ. Η ηλεκτρονική επαλήθευση, μάλλον η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τροπολογία 80, πέρα της ψηφοφορίας και απορρίπτεται 9 με 13. Τροπολογία 81 υπέρ. Εποχές ε, εγκρίνεται. Τροπολογία 82 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 84 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 85 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση για το 85 άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 12 υπέρ 10 κατά. Τροπολογία 17 και 86 ταυτόσιμες από κοινού υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 87 υπέρ κατά. ηλεκτρονική επαλήθευση για το 87. Πέρας και εγκρίνεται. 14 υπέρ 8 κατά. Ο 18 δεν θα ψηφιστεί. Τροπολογία 88 υπέρ. Υπέρ. Κατά. Α, ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 88. Εγκρίνεται 19 και 89 από κοινού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 20 και 19 υπέρ κατά, και 90 συγγνώμη υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται 91 ε, ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 91 πέρας εγκρίνεται 12 με 10 92 υπέρ η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 92 άρχεται η ψηφοφορία πέρας 12 με 10 εγκρίνεται, τροπολογίες 21 και 93 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 94 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 95 υπέρ, ε, ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 95 άρχεται η ψηφοφορία. Απορρίπτεται 10 υπέρ 12 κατά. Τροπολογία 96 υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται 97 υπέρ κατά ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 97 άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 14 υπέρ 8 κατά τροπολογία 22 υπέρ 22 υπέρ κατά ε, ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 22 άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 12 υπέρ 10 κατά τροπολογία 98 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 99 υπέρ ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 99 άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται 9 υπέρ 13 κατά δεν λειτουργεί ε, ναι ούτως ή άλλως καταγράφηκε η ψηφοφορία σας ε, τροπολογία 100, 100 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 101 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 102 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 104, 104 υπέρ κατά ε, να επαληθεύσουμε την 104 με ηλεκτρονική ψηφοφορία, πέρας της ψηφοφορίας και απορρίπτεται 10 υπέρ 11 κατά. Η 107 ήταν ταυτόσημη, επομένως περνάμε στην 25 και την 105 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 106 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 108 υπέρ η ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 108, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας πρέπει δύο ακόμα να ψηφίσουν, δεν θέλουν να ψηφίσουν, εν πάση περιπτώσει εγώ κλείνω την ψηφοφορία. Και εγκρίνεται 12 υπέρ 9 κατά. Τροπολογία 28 στις αιτιολογικές σκέψεις υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 38 υπέρ εδώ δεν έχουμε ενιαία γραμμή, άρα ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τροπολογία 38. Ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία 38 πέρα της ψηφοφορίας και εγκρίνεται 12 ψήφοι υπέρ, 10 κατά. Τροπολογία 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 40 υπέρ κατά. Μπάρμπαρα, όταν δεν σηκώνει το χέρι σου απέχεις. 40 ε, εγκρίνεται η 40. 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 3 και 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, τελική ε, ψήφος διονομαστική, ψηφοφορία διονομαστικής εκκλήσεως, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 20 υπέρ 2 κατά εγκρίνεται λοιπόν. Ε, δεν φαίνεται να έχουμε κάτι άλλο στην ημερήσια διάταξη, άρα μάλλον ε, ολοκληρώθηκε η πρωινή μας συνεδρίαση. Αγαπητοί συνάδελφοι, ε, παρακαλώ τους συντονιστές 5-10 λεπτά να ε, κάνουμε μία πολύ σύντομη συνεδρίαση τώρα, έτσι ώστε να μην κάνουμε την συνάντηση αυτή μετά τις 12.30. Εάν μπορείτε οι συντονιστές να παραμείνετε, ε, θα κάνουμε τη, συνάντηση, τη συνεδρίας των συντονιστών.